Σήμερα το βράδυ είναι η προσχώρηση ε, του Εκουαντόρ, του Περού και της Κολομβίας στην Εμπορική Συμφωνία. Και θέλω να δώσω και το λόγο και πάλι στην Επίτροπο κυρία Μάλφρυ. Να δω λιγάκι, μισό λεπτό βρήκα τα χαρτιά μου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, χαιρετίζουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που αφορά στην Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Περού και προσφόρηση του Εκουαντόρ. Αυτό ε, συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, το Περού και την Κολομβία και είναι άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός στην προσπάθειά μας για να σταθροποιήσουμε τη σχέση μας στη Λατινική Αμερική. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτή η συμφωνία θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές θα μας δώσει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσουμε τις παραδοσιακές ροές, να ενισχύσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις και στις δύο πλευρές. Επίσης πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα είναι οικονομική στήριξη για τον Ισημερινό, θα βοηθήσουν στο να εξαλειφθεί η φτώχεια και οι ανισότητες, που βεβαίως και υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Το ε, πρωτόκολλο της ε, προσχώρησης ε, έχει πολλά φιλόδοξα στοιχεία όπως αυτό που συνήθει και με την Κολομβία και το Περού. Βεβαίως και λαμβάνουν υπόψη οι διαφορές της οικονομικής ανάπτυξης στο Εκουαντό, στον Ισημερινό με και βεβαίως υπάρχουν και κάποια, κάποιες ειδικές προϋποθέσεις που ζήτησε ο Ισημερινός. Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η συμφωνία από του χρόνου ο σημερινός δεν θα έχει πλέον προνομιούχο μεταχείριση. Και γι' αυτό, ε, εάν υπάρχει έγκαιρη προσχώρηση, αυτό θα συνεπάγεται μακροχρόνια σταθερότητα και ε, συγκεκριμένες προβλέψεις για το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις. Όπως συζητήσαμε και προηγουμένως και εξήγησα και στην εμπορική μας στρατηγική θα αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία έτσι ώστε οι διατάξεις για το εμπόριο, ε, την εφόρο ανάπτυξη να εφαρμόνται σωστά ε, μέσα από την αναπτυξιακή συνεργασία. Ο σημερινός και το βλέπετε αυτό, έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να ασχοληθεί με το εμπόριο και με την αηφόρο ανάπτυξη. Και έχει συμφωνήσει να υπογράψει όλες τις διατάξεις των κεφαλαίων αηφόρο ανάπτυξης. Αυτό θα μας βοηθήσει να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές, όπως και σε άλλες περιπτώσεις η συνεργασία με εσά θα είναι καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική εφαρμογή τη συμφωνία, κυρίω για το κεφάλαιο τη αηφόρου ανάπτυξη. Για να γίνουν όλα αυτά, χρειαζόμαστε την αφοσίωσή σα, την συνεισφορά σα. Το ε, ψήφισμα αυτό νομίζουμε ότι εκφράζει την ε, συνεισφορά σα. Λάβαμε υπόψη μα αυτό που ζητάτε ε, να ενημερώνεστε για την εισαγωγή από μπανάνες από τον Ισημερινό και μπορώ να σας διασφαλίσω ότι ο αυστηρός έλεγχος εισαγωγών μπανάνας ε, αποδεικνύεται μέχρι τώρα αποτελεσματικός. Το ψήφισμα είναι καθοριστική σημασίας για την προσχώρηση του Ισημερινού. Βεβαίως δεν τελειώνει και η συζήτηση. Θα συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η συμφωνία ε, και μέχρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μπορεί να λάβει σοβαρά υπόψη της όπως και το διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ για το ψήφισμα και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, μέχρι να τεθεί σε ισχύ. Ο κύριος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Τον Ιούλιο πέρσι ε, εστέφθηκαν από επιτυχία οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ε, Ισημερινού Κολομβίας και Περού και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ θετικό και για τα δύο μέρη, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ισημερινός ζήτησε να ενταχθεί στις διαπραγματεύσεις που είχε εγκαταλείψει το 2009. Γι' αυτό και μετά από ρήτρα διασφάλισης ε, ε, καταφέραμε να εντάξουμε και τον Ισημερινό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτς για την ε, πολύ καλή έκβαση των διαπραγματεύσεων. Το ΕΛΚ έχει υποβάλει τροπολογίες στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για να εμπλουτίσουμε το κείμενο και να δείξουμε και την υποστήριξή μας προς τον Ισημερινό. Αυτό αντικατοπτρίζεται και από το τελικό κείμενο έτσι ώστε να προωθήσουμε την, το εμπόριο από όλες τις πλευρές και να καταπολεμήσουμε και τις ανισότητες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχει σημασία να λάβουμε υπόψη και το καθεστώς γενικευμένων προτιμήσεων πλάς. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στις 13 Ιουνίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν συμφωνήσει τελικά ε, όρισε έναν οδικό χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ε, δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Έτσι ώστε να συμμετάσχουν και οι τρεις χώρες στη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Λάγκε για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πράγματι εμείς ε, χαιρετίζουμε την προσχώρηση του σημερινού στη συμφωνία διότι ε, θέλαμε να έχουμε μια συμφωνία με τις Άντις διότι η ενσωμάτωση σε περιφερειακό επίπεδο είναι καθοριστικό στοιχείο της πολιτικής μας έναντι των χωρών στη Λατινική Αμερική. Με το ψηφίσμα λοιπόν αυτό ε, Είχαμε, επιτύχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Σόλτ, με τον κύριο Φίσα και με όλου του άλλου ε, εμπλεκόμενου. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σωστή είναι λοιπόν η κατεύθυνση. Θέλουμε να οργανώσουμε την ε, ένταξη αλλά και την εφαρμογή. Και γι' αυτό το λόγο παραπέμπουμε στον οδικό χάρτη που επιτύχαμε στην Κολομβία και στο Περού τότε με τον Μάριο Ντάβιτ και με την ταπεινότητά μου. Ε, εμείς λοιπόν διαπραγματευτήκαμε αυτό τον χάρτη πορείας με τις ε, κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Κύριε Πρόεδρε, σημαντικές δεν είναι μόνο οι αποφάσεις αλλά και η εφαρμογή των αποφάσεων. Επίσης ε, σημαντικό είναι το τι γίνεται με τους εργαζόμενους, ε, με το περιβάλλον από κοινού. Πρέπει να τα καθορίσουμε αυτά για να επιτύχουμε βελτιώσεις. Κατόπιν τούτου το, ο Ισημερινός καλείται να ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση όπως και η Κολομβία και το Περού ε, για να επιτευχθεί πρόοδος κυρίως όσον αφορά το θέμα των επιθεωρητών εργασίας διότι ε, δεν έχει ακόμα υπογραφεί η Συμφωνία Υπαριθμών 29 των Ηνωμένων Εθνών. Άρα δηλαδή από κοινού πρέπει να προσπαθήσουμε και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας. Κυρία Μπιλμπάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη υποστήριξή μας για την προσχώρηση του Εκουαδό στη συνθήκη ελευθέρω εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία έχει υποφελθεί από το 2013 η Κολομβία και το Περού. Έχουν χαθεί δύο χρόνια και ελπίζω ότι για το Εκουαδόρ θα είναι τα ίδια τα ωφέλη τα οποία θα προσποριστεί από τη συμφωνία αυτή όπω η Κολομβία και το Περού. Μόνο στην Κολομβία υπήρξε όφελο για 4 εκατομμύρια οικογενειών γεωργών που ήταν να αυξάνονται κατά 21% οι εξαγωγέ του η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριο αποδέκτη εξαγωγών από το Εκουαδόρ. Το 2014 οι πωλήσει στην αγορά μα έφτασαν τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ευρώ με 400 εκατομμύρια εμπορικό πλεόνασμα για το Εκουαδόρ. Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν και πάρα πολλέ επιχειρήσει οι οποίε έχουν επωφεληθεί από αυτέ τι εμπορικέ ροέ. Μπορούν έτσι να βελτιώσουν τι ε, ανταλλαγέ για άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ στο άμεσο μέλλον. Έτσι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα θαυμάσιο εργαλείο για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ειρήνη, στη σταθερότητα και την πρόοδο στην περιοχή αυτή. Με τον τρόπο αυτό έχουμε ανάπτυξη, έχουμε οικονομική μεγέθυνση και εγγύηση σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Οδηγεί σε κοινωνική σταθερότητα και <clears throat> δικαιοσύνη για μια περιοχή που είναι νευραλική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία έχει σημαντικό χαρακτήρα ως περιοχή οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, Πολλοί πολίτες, πολίτες της χώρας αυτής έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέλει να εξάρει τη σημασία αυτών των συμφωνιών που δίνουν απτά αποτελέσματα σε χιλιάδες οικογενειών και εργαζομένων που έχουν την ευκαιρία να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους σε εμπορικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ελπίζω και η Βολιβία θα, θα συνταχθεί σε αυτή τη συμφωνία η οποία θα είναι ωφέλιμη για όλη την κοινότητα των άνδρων. Είναι μια λοιπόν πολύ σημαντική ευρωπαϊκή συμβολή στην ειρήνη, την δικαιοσύνη και την παγκοσμία ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς κυρία Πίτροπε η ομάδα μας θα υποστηρίξει μαζί σα την ε, προσπάθεια αυτή της Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η κυβέρνηση του Εκουαδόρ έχει αποφασίσει να ακολουθήσει την Κολομβία και το Περού και να μπει στην συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε εξαναγκαστικά γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μην έχει να αντιμετωπίσει ε, αθέμητο ανταγωνισμό από τους δύο γειτονέ τους. Το Εκουαδόρ θα έπρεπε να έχει τη δική του ε, συμφωνία όπως είχε προταθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν ήθελε να έχει μια εταιρική σχέση με χώρες αυτές θα έπρεπε να δίνει και πολύ μεγαλύτερη σημασία στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη χώρα αυτή. Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμφωνία με την Κολομβία και το Περού, όπως ξέρετε, καθυστέρησε για πολύ καιρό και ήταν ιδιαίτερα επίμαχη και έγινε δεκτή μονάχα υπό την προπόθεση ότι θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα σε κοινωνικό επίπεδο και για την προστασία του περιβάλλοντο και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Αυτοί είναι στόχοι για του οποίου εμεί εμείς έχουμε. Ε, έχει αγωνιστεί η κυβέρνηση του Εκουαδόρ. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας. Η ε, προσχώρηση του Εκουαδόρ σε αυτή τη συνθήκη είναι μια πάρα πολύ σημαντική χρονική στιγμή για την ίδια τη χώρα, αλλά επίσης για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες αυτές πάντα θα περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική δικαιοσύνη σε όλες τις χώρες της περιοχής. Τα πρώτα δείγματα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει στις συμφωνίες με τις δύο άλλες χώρες προς την κατεύθυνση αυτή που είχε διαγραφεί. Θα πρέπει λοιπόν επίσης και για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και όχι μονάχα για την υπογραφή της να ασχοληθούμε και να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουμε το σωστό τρόπο. Με το ψήφισμα αυτό εγώ τονίζω την ανάγκη εμείς να επομιστούμε τις ευθύνε μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να καταδείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι να ε, εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτού του, αυτής της συμφωνίας όταν πράγματι είναι προς όφελος των πληθυσμών και των δύο περιοχών. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους σκιώδεις εισηγητές τη ομάδα μου για το γεγονό ότι καταλήξαμε σε ένα ψήφισμα το οποίο θεωρώ ικανοποιητικό. Ευχαριστώ. Ο κ. Μάτο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η ένταξη του σημερινού στην συμφωνία με Πέρου και Κολομβία θα ανοίξει πολλές ευκαιρίες για όλες τις πλευρές, αλλά τα ωφέλη θα επιτευχθούν μόνο αν εργαστούμε ε, σκληρά και τηρηθούν ε, στο ακέραιο όλες οι προϋποθέσεις. Ε, θα ήθελα να αναφέρω, ε, λόγω και της παραγωγής μπανάνας, ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες απειλές για τον τομέα της μπανάνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα μπορούσε να υπάρξει ανεξέλεγκτη εισαγωγή μπανανών από τον Ισημερινό. Είναι μεγαλύτερο εξαγωγέα ε, μπανανών η χώρα του Ισημερινού και ακριβώς ε, ε, όσο μειώνονται οι δασμοί αυξάνονται οι εξαγωγέ. Είχαμε μιλήσει για δασμούς της τάξης των 114 ευρώ τον τόνο και έχουμε πει ότι θα πέσει 74 ε, σε λίγα χρόνια και θα το κάνουμε. Απλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η αντιστάθμιση στους κοινοτικού παραγωγούς, αποζημιώσεις γιατί μπορεί να πληγούν και δεύτερον θα πρέπει με τη δέωση επιμέλεια να εφαρμοστεί ρήτρα εξασφάλισης σε περίπτωση που ε, υπερβούν οι ε, παραγωγοί του σημερινού αυτές ποσοστός προκαλώντας ζημία στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ναι, να ενταχθεί σε αυτή τη συμφωνία ο σημερινός και ναι, να αναπτυχθεί η χώρα όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα και ιδίω ε, σε βάρος των παραγωγών μπανάνας από τα Κανάρια νησιά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτή η ρήτρα διασφάλισης που είπα. Θα πρέπει όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε και να τα τηρήσουμε αλλιώς θα πρέπει πρέπει αυτόματα να ενεργοποιείται ο μηχανισμός όταν υπάρχει υπέρβαση των ποσοστώσεων. Αυτό ε, θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Δεν θα πρέπει να έχει διαφορετική μεταχείριση ο σημερινός ε, καλύτερη από το ε, Περού και την Κολομβία. Αυτή τη ρήτρα διασφάλισης πρέπει να τη θέσετε σε ισχύ και να μην ξεχάσετε την άλλη πλευρά, να μην στρέψετε αλλού το βλέμμα ξεχνώντας τις οικογένειες που ζουν από την Πανάνα στις, στα Κανάρια νησιά και σε άλλες εξόγως από περιφέρειες. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό, κύριος Χαουρέγγι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε ότι η Λατινική Αμερική είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση από εμπορική έποψη. Ιδίω όπως και άλλοι σημαντικοί εταίροι σε παγκόσμιο επίπεδο, όπω η Κίνα αυτή τη στιγμή, διεκδικούν αυτή την αγορά. Για την κοινότητα των χωρών των Άνδεων, του Εκουαδόρ είναι μια πάρα πολύ σημαντική χώρα. Πιστεύω επίση ότι για τον πολιτικό περίγυρο της λεγόμενης κοινότητας των χωρών των Άνδεων, το Εκουαδόρ και ο πρόεδρος του Κορέα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι είναι πολιτική επιταγή και εμπορική επιταγή το να μπορέσει να γίνει αυτή η συμφωνία και συμφωνώ με όλους αυτούς οι οποίοι το διεκδίκησαν εδώ. Το Εκουαδόρ ίσως έκανε σφάλμα όταν αποφάσισε πριν από δύο χρόνια να μην ακολουθήσει την Κολομβία και το Περού. Τώρα όμω είναι φανερό ότι μα δείχνει με κατηγορηματικό και σαφή τρόπο ότι θέλησή του σε πολιτικό επίπεδο να μπορέσει να συνταχθεί με τι άλλε δύο χώρε σε αυτή τη συμφωνία και μα φέρνει και επίση το άγχο που νιώθει σε οικονομικό επίπεδο ότι είναι απαραίτητο αυτή η συμφωνία το ταχύτερο δυνατό να μπορέσει να συναυθεί για να εξασφαλιστεί το μέλλον των εξαγωγών του. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει τα απαραίτητα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο που να έχει να κάνει με ε, αηφόρο ανάπτυξη, αηφόρο εμπόριο και ανθρώπινα δικαιώματα που να αντιτίθεται σε μια τέτοια συμφωνία. Είναι μια πολύ σημαντική εμπορική συμφωνία που θα έχει σημαντική πολιτική επίπτωση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει την Κομισιόν και να περατώσει τι διαπραγματεύσει και να ακολουθήσει έτσι το Ακουαδό, την Κολομβία αλλά και το Περού. Σα ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ροντρίγκε Πινιέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον συντάκτη του ψηφίσματο, γιατί ήταν ανοιχτό στο διάλογο, στη συνένεση και έκανε και εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα να τονίσω και εγώ την ε, στεναρή υποστήριξη ε, της ισπανικής αντιπροσωπείας ε, της σοσιαλιστική ομάδα. Στις δεσμεύσεις για διατήρηση των πολιτικών σχέσεων με τον Ισημερινό. Χαιρόμαστε και συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά της που θα επιτρέψει την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία με Κολομβία και Περού. Θεωρούμε όμως ότι αυτή η συμφωνία, όπως έλεγε προηγουμένως ο κύριος Χάουρεγγι, αυτή η συμφωνία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μέσα στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψουν στη χώρα του σημερινού να αποφεληθεί όλων των ε, πλεονεκτημάτων αυτή τη συμφωνία. Όμω, για την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξίσου ε, μεγάλη σημασία, για, μάλλον με την εμπορική πολιτική, έχει και η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ ενό κεφαλαίου για βιώσιμη εφόρα ανάπτυξη με σαφεί όρου και προποθέσει ό,τι αφορά εργασιακά δικαιώματα, συνδικαλιστικέ ελευθερίε, καταπολέμηση τη παιδική εργασία, προάσπιση τη ισότητα των δύο φύλων, προστασία των αυτόχθονων πληθυσμών και για μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ελπίζουμε έτσι να γίνει και θα παρακολουθούμε την ε, συμφωνία προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ένταξη του Ισημερινού στη συμφωνία με το Περού και την Κολομβία είναι ένα περαιτέρω βήμα για τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική. Αναμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι διευρύνεται η εμβέλεια ε, της συμφωνίας αυτής σε κοινωνικούς τομείς και σε περιβαλλοντικούς και οικονομικούς. Θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις για την βελτίωση των συνθήκων ζωής και εργασίας των πολιτών του Ισημερινού. Πέρα από τις ειδικέ σχέσεις θα έλεγα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στα πλαίσια του συστήματος γενικών προτιμήσεων βλέπουμε ότι η Λατινική Αμερική παραμένει για οικονομικούς και πολιτιστικούς λόγους μια στρατηγική περιοχή, μια περιοχή καλύτερα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αντίστοιχες ρυθμίσεις με το σύνολο της περιοχής Μερκοσούρ ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι η συμμετοχή ε, του Ισημερινού στη συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την Κολομβία και το Περού είναι ένα θετικό βήμα. Είναι κάτι το οποίο πρόκειται να ωφελήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εγώ πήρα μέρος στην διαδικασία αυτή, την παρακολούθησα στα πλαίσια του Eurolat και ήμουν πάντα υπέρ της εμβάθυνσης της συνεργασίας με τη Λινική Αμερική. Νομίζω ότι ο Ισημερινός είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας χώρας η οποία προοδεύει. Συμφωνίες τέτοιου είδους με τους εμπορικούς εταίρους μας έχουν σημαντική θα έλεγα διάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τόλμησε στη σύγχρονη εποχή να προχωρήσει θαραλέα στη διαγραφή του εξωτερικού χρέους της χώρας προς τρίτους και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. σήμερα συζητούμε την ένταξη του ισημερινού στην εμπορική συμφωνία της ευρωπαϊκής ένωσης με το περού και την κολομβία. για να είναι όμως επωφελής η συμφωνία για τον ισημερινό θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια προκειμένου η απελευθέρωση του εμπορίου να αποβεί υπέρ του λαού του ισημερινού και όχι των πολυεθνικών αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη τοπική απασχόλησης των εργασιακών δικαιωμάτων και της αγροτικής οικονομίας και αυτό δεν μπορεί να γίνει με εμπορικές συμφωνίες που προωθούν μια πλήρη και άνευ όρων απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. απαιτείται λοιπόν ένα δίκτυ προστασία για τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε και για του φτωχού και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί αντιστάθμισης των κοινωνικών επιπτώσεων από το άνοιγμα της αγοράς του ισημερινού στις επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. Ο κύριος Γιακοβτσίτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη συμφωνία η οποία θα υπογραφεί με το Περού, την Κολομβία και τον Ισημερινό αποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Πολύ σωστά λοιπόν υπόθηκε ότι είναι θετική η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με αυτές τις χώρες γιατί έτσι αποδεικνύεται έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για αυτές. Αυτό όμως είναι και επιβεβαίωση της μεγάλης σημασίας την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκόσμια εμπορική σκηνή. Και φυσικά θα πρέπει εδώ να βοηθήσουμε και τους ηθαγενείς πληθυσμούς του Ισημερινού που εμπλέκονται στη γεωργική παραγωγή χωρίς να ε, βλάψουμε φυσικά τους παραγωγούς ε, φρούτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στις νήσους Καναρίους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είπατε πολλοί από εσά, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα θέματα συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολοβίας Περού και Εκουεδόρη. Η συμφωνία με την Κολοβία και το Περού είναι μια καλή συμφωνία όπως ελέγχθη <clears throat> και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και το Εκουαδόρ, για, το Εκουαδόρ. Υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί για το Εκουαδόρ, λαμβάνοντα υπόψη τι διαφορέ των οικονομιών των τριών χωρών. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι μηχανισμοί για να του επιτρέψουν να αναπτύξουν περαιτέρω την οικονομία του, αλλά συγχρόνω να αντιμετωπίσουν και τα κοινωνικά θέματα τα οποία εμπλέκονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά επίση και για την περιφερειακή ολοκλήρωση του επίπεδου των χωρών αυτών. Θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων και τη αηφόρου αναπτύξεως και άλλα θέματα. Η δεύτερη έκθεση για το Περού και την Κολομβία είναι στα τελικά της στάδια. Θα σας αποσταλεί συντόμως. <clears throat> για τις μπανάνες. Ε, άκουσα τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένοι από εσά. Έχουμε ένα μηχανισμό σταθεροποίησης και παρακολουθούμε προσεκτικά την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού ώστε να ε, παρακολουθούμε την κατάσταση, θα σας κρατούμε ενήμερος και φυσικά έχει και το Εκουαδόρ ένα μηχανισμό διασφάλισης. Θα, θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός αυτός καλύπτει και τις ανάγκες του Εκουαδόρ και θα δίνουμε τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα για τη γενική υποστήριξη που έχετε εκδηλώσει. Εγώ προσβλέπω σε μια στεναρή υποστήριξή σας σε σχέση με το ψήφισμα το οποίο θα έρθει αύριο σε ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Το έχουμε αναδειφθεί προσεκτικά, έχουμε μελετήσει και τις τροπολογίες και πιστεύουμε ότι το ψήφισμα αυτό θα μπορέσει να μας βοηθήσει ιδιαίτερα για να συμπληρώσουμε τον αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε.